Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann eröffne ich wieder die Sitzung. τη συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφοι, στο σημείο 17 Okay. Punkt äh, siebzehn ist der Austausch. Ανταλλαγή λοιπόν απόψεων στο σημείο 17 με τον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Την πρέσβη, την κυρία Γιάνγκ Λί. Δεν τίποτα θέμα. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος συμπορικός εταίρος και έτσι σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα εμπορικών ε, κινήτρων και να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτά. Για μια επενδυτική συμφωνία ίσως και κάτι παραπάνω σε κάθε περίπτωση. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την ε, ασφάλεια και την κατάργηση των περιορισμών στο εμπόριο και στις επενδύσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερως κυρία Πρέσβη που βρίσκεστε μαζί μας. Έχουμε διερμηνία και από τα Κινέζικα. Μπορείτε να μιλήσετε λοιπόν κινέζικα και να ακούτε κινέζικα στο κανάλι 22. Και θα σας δώσω λοιπόν το λόγο παρά αυτά. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπέρντ Λάγκε, πρόεδρε της ΣΥΝΤΑ, κύριε Λίλο Βίνκλερ, πρόεδρε της ε, ομάδας εποπτείας για την Κίνα και κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας μιλήσω σήμερα. Πριν αρχίσω τα σοβαρά θέματα θα ήθελα να σας στείλω ευχές σε όλα σας τα μέλη διότι πολλά χρόνια από τότε που άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας η ΙΝΤΑ έχει παίξει σοβαρότατο και απαραίτητο ρόλο για την προώθηση εμπορικών δεσμών μεταξύ Κίνας και Ένωσης και εκτιμούμε ιδιαίτερα όλη την αφοσίωση και τη συμβολή σας. Η Κίνα και οι σχέσεις της με την Ένωση είναι γνωστές σε εσά. Αλλά λόγω του περιορισμού του χρόνου θα ήθελα να περιοριστώ σήμερα σε τρία θέματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Πρώτον, η σημασία της Κίνας για την Ένωση, δεύτερον η μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας και τρίτον περαιτέρω επέκταση των εμπορικών δεσμών Κίνας και Ένωσης. Η κινέζικη οικονομία έφτασε σε καινούργια φάση. δηλαδή, μειώνει λίγο την ταχύτητα ανάπτυξής της από ένα πρότυπο που βασιζόταν στην ταχύτητα και την ποσότητα σε ένα πιο εντατικό πρότυπο με βάση την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα. Από την έμφαση στην επένδυση σε εργοστάσια, έμφαση τώρα στην καινοτομία. Καθώς η οικονομία συνεχίζει να αυξάνεται και να αναπτύσσεται σε ποσοστό περίπου 7% δημιουργείται μία ορμή, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης στο παρελθόν ήταν διψήφιος. Η κινέζικη οικονομία λοιπόν είναι πολύ ανθεκτική και έχει μεγάλες δυνατότητες, μας αφήνει χώρο για να εφαρμόσουμε πολλά εργαλεία πολιτικής με μεγαλύτερη δημιουργικότητα. Όπως προβλέπεται και από μία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, με αυτή την αλλαγή της αναπτυξιακής στρατηγικής και την προσαρμογή στις νέες προκλήσεις, η Κίνα είναι σε καλή θέση για να γίνει μία σύγχρονη κοινωνία υψηλών εισοδημάτων μέχρι το 30. Είμαστε βέβαιοι ότι η Κίνα θα μετατραπεί σε μία ευημερούσα κοινωνία μέχρι το 20 ήδη και με ισχυρή δημοκρατία και πολιτιστικά προοδευμένη χώρα μέχρι τα μέσα του αιώνα. Η κινέζικη οικονομία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ανάπτυξη, πιο πολύπλοκη κατανομή εργασίας και καλύτερες δομές που ελκύουν και άλλους επενδυτές στην Κίνα. Χάρη στις μεταρρυθμίσεις μας οι εμπορικές σχέσεις με την Ένωση έδειξαν μεγάλη αύξηση από 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 1975 σε 615 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Σημαντικότατη αύξηση 250-2.500% όχι 25.000%. Και η Κίνα είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος της Ένωσης. Κάθε μέρα η Κίνα και η Ευρώπη συναλλάσσονται σε πολύ υψηλά ποσά, σαν δισεκατομμύρια. Η... Το πρόγραμμα της Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση θα ωφεληθεί και από την καινούργια φάση της Κίνας η εκβιομηχάνηση, οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ο εξυγχρονισμός της γεωργίας, η πράσινη ανάπτυξη και η εισαγωγή, τεράστιες εισαγωγές καθώς και επενδύσεις θα δημιουργήσουν περισσότερες δυνατότητες εμπορίου, συναλλαγών και συνεργασίας και για άλλες χώρες και περιφέρειες. Και οπωσδήποτε θα διευκολυνθεί έτσι η αναθέρμανση των δομικών μεταρρυθμίσεων της Ένωσης για να... και θα υπάρχουν συγκλινόμενα συμφέροντα μεταξύ των δύο χωρών. Δεύτερον, η μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας πεπισμένοι ότι οι μεταρρυθμίσεις και το άνοιγμα είναι ζωτικά για την ανάπτυξη, η Κίνα εμβαθύνει τις μεταρρυθμίσεις της και τις δομικές προσαρμογές της. Μεταξύ άλλων, αυξάνει τις προσπάθειές της να απλοποιήσει την δημόσια διοίκηση και δίνει περισσότερες δικαιοδοσίες σε αποκεντρωμένες δομές για να μειωθούν οι φραγμοί και η αναποτελεσματικότητα. Επίσης, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και των κρατικών επιχειρήσεων και του κρατικού κεφαλαίου. Συνεχίζει να ανοίγει την πολιτική της για περισσότερη φιλελευθεροποίηση και διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων ενώ παράλληλα κρατάει τις εξαγωγές σταθερές αν και αυξάνει τις εισαγωγές. Πέρυσι οι ξένες επενδύσεις στην Κίνα έφτασαν τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια καθιστώντας την Κίνα την πρώτη χώρα για επενδύσεις από ξένους. Ενώ οι επενδύσεις της Κίνας στο εξωτερικό είναι περίπου ισοδύναμες με αυτές. 150 μάλλον δισεκατομμύρια. Ο πρόεδρος Σιν κατέστησε απολύτως σαφές ότι η Κίνα θα ανοιχτεί ακόμη περισσότερο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν θα αλλάξει η πολιτική ενθάρρυνση των ξένων επενδύσεων και τα δικαιώματα των επενδυτών, οι ξένες εταιρείες θα προστατεύονται και θα χορηγούνται καλύτερες υπηρεσίες με στόχο να δημιουργηθεί μια καινούργια ανοιχτή οικονομία. Εξυγχρονίζουμε και τις δομές του εξωτερικού μας εμπορίου και του εμπορίου υπηρεσιών με πιο ενεργή πολιτική και χρήση της προωθημένης τεχνολογίας και εγκαταστάσεων. Επίσης, είμαστε πιο ενεργοί στη χρήση ξένων κεφαλαίων για τη δημιουργία μιας σταθερής δίκαιας διαφανούς και προβλέψιμου περιβάλλοντος, επιχειρησιακού περιβάλλοντος με το καινούριο νομοσχέδιο για τις ξένες επενδύσεις και με την αναθεώρηση του καταλόγου επιχειρήσεων που επενδύουν με στόχο να βελτιωθεί το σύστημα διαχείρισης των ξένων επενδύσεων Τελεία. Ε, εξίσου σημαντικό είναι ότι η Κίνα έχει αρχίσει να εφαρμόζει ένα νέο σύστημα για την εξέταση και αδειοδότηση των ξένων επενδύσεων με βάση μια τράπεζα δεδομένων. Για να δημιουργηθεί αυτό το καινούργιο περιβάλλον και το άνοιγμα, η Κίνα συνεργάζεται και με άλλες χώρες για να αναπτυχθεί η οικονομική ζώνη του δρόμου του μεταξιού. Επίσης αναπτύσσει στη Σανγκάη, στην Κουαντούγκ, στο Κέντζιν και στο Φουτζιάν πειραματικά προγράμματα για την εφαρμογή ενός νέου προτύπου ή μοντέλου για τις επενδύσεις με νέο σύστημα αδειοδοτήσεων και βελτίωση της νομοθεσίας. Όπως δείχνουν και τα οικονομικά μας αποτελέσματα πέρυσι, ο νέος γύρος αυτός των μεταρρυθμίσεων και του ανοίγματο κατέληξε στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και θα συνεχίσει αυτό. Τρίτον, περαιτέρω επέκταση των σχέσεων, των εμπορικών σχέσεων Κίνας Ένωσης. Τις περασμένες τέσσερις δεκαετίες οι σχέσεις αυτές ήταν ενδεικτικές μπορεί να είχαν διαφορετική ιστορία, πολιτισμό, ιδεολογία και κοινωνικά συστήματα οι χώρες, αλλά εφόσον είναι διατεθειμένες να σεβαστούν η μία την άλλη και να συναλλαχθούν ε, ισότιμα, μπορούν να έχουν αμοιβαία ωφέλη. και μια στρατηγική εταιρική σχέση. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι και η Κίνα και η Ένωση εκμεταλλεύονται πλήρως την 40η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων Ένωσης Κίνας που γιορτάζουμε φέτος. Για να συνεχιστεί ο ψηλός ρυθμός επισκέψεων ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Σούλτς πρόσφατα πήγε στην Κίνα και η, πάτη κυρία Μογκερίνη πήγε επίση στο Πεκίνο για να συμπροεδρεύσει με τον Γιάνν Κετσού την τον πέμπτο διάλογο υψηλού επίπεδου Κίνας Ένωσης. Και η, σίγουρα εν καιρό το δέοντι θα γίνει εδώ στις Βρυξέλλες και η 7η κοινή διάσκεψη Κίνας Ένωσης για αξιολόγηση των τιμερών σχέσεων και για καθορισμό της μελλοντική πορείας. Η διάσκεψη αυτή θα ακολουθηθεί από νέους γύρους διαλόγων υψηλού επίπεδου και εμπορικών και πολιτιστικών. Για να ανταποκριθούμε λοιπόν στις προτεραιότητες των προγραμμάτων μας και να διασφαλίσουμε ότι οι οικονομίες μας θα παραμείνουν πρωτοπόρες παγκόσμια, η Κίνα και η Ένωση συνεργάζονται για να εφαρμόσουν τους κοινού στόχους 2020 Κίνας Ένωσης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην διαπραγμάτευση για μια συμφωνία διμερών επενδύσεων η οποία πρέπει να επιταχυνθεί πράγμα το οποίο δείχνει το κοινό μας όραμα για την εφαρμογή ενός κοινού νομικού πλαισίου ώστε να υπάρχει προβλέψιμη μακροπρόθεσμη πρόσβαση στις δύο αγορές και για ισχυρή προστασία των επενδυτών και των επενδύσεών των. Από τα τέλη του 2013 η Κίνα και η Ένωση οργάνωσαν πέντε γύρους διαπραγματεύσεων επικοδομητικών τον πέμπτο γύρο των διαπραγματεύσεων που τελείωσε πριν από μερικές εβδομάδες οι δύο πλευρές συνέχισαν να ανταλλάσσουν απόψεις για το προτινόμενο κείμενο θέτοντας έτσι τα θεμέλια για τις μελλοντικές τους διαπραγματεύσεις. Για να υπάρξει η πρόοδος που χρειάζεται για κοινή ευημερία, η Κίνα επιταχύνει την εφαρμογή της στρατηγικής ενός χώρου ελευθέρων συναλλαγών και με την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων και με την Αυστραλία θα θέσουμε θεμέλια και για μια περιφερειακή οικονομική εταιρική σχέση με την Ιαπωνία και την Αυστραλία που είναι για μας προτεραιότητες. Ελπίζουμε η Κίνα και η Ένωση να συνάψουν και μία τέτοια εμπορική συμφωνία μεταξύ τους, FTA, Foreign Trade Agreement. Να κάνουν δηλαδή καταρχήν κοινέ ε, μελέτες για τα προοπτικές μιας τέτοιας συμφωνίας που θα είναι μια κατάσταση win-win και για την Κίνα και για την Ένωση. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η Κίνα και η Ένωση συνεργάζονται για να βρουν τρόπους διευκόλυνσης των συναλλαγών και των ανταλλαγών για τους πολίτες της Ένωσης και της Κοινός, όπως διευκόλυνση των θεωρήσεων για τη δημιουργία συνθήκων, καλύτερων συνθήκων και εμπορικών, αλλά και γενικότερα επιχειρηματικών με στόχο την αποτελεσματικότητα, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της συνεργασίας αυτής είναι η διαχείριση των το, ορισμένων τοξικών ουσιών όπου η Κίνα και η Ένωση έλυσαν το πρόβλημα, α, κρεμών προβλημάτων μάλλον, όπως των ηλιακών και των βολταϊκών και λόγω του μεγέθους, του ύψους των συναλλαγών Κίνας Ένωσης ήταν αναπόφευκτο να υπάρξουν και μερικές τριβές εμπορικές, μεγάλες ή μικρές. Τελείως φυσικό. Το θέμα όμως είναι η πολιτική θέληση και της Κίνας και της Ένωσης να κρατήσουν τα μακροπρόθεσμα κοινά του συμφέροντα και να λύσουν με επικοδομητικό τρόπο μέσω διαλόγου οποιασδήποτε τριβές και διαφωνίες με αμοιβαία υποφελή τρόπο πιστεύουμε ότι οι σχέσεις Κίνας-Ένωσης είναι όριμες, ανθεκτικές και αρκετά σταθερές και δυνατές ώστε να υπομείνουν επιτυχώς οποιασδήποτε δοκιμασίες. Και τέλος, στον με βάση τον ΠΟΕ η Κίνα είναι έτοιμη να βελτιώσει το συντονισμό και τη συνεργασία με την Ένωση και να προωθήσει τον γύρο της Δόχας καθώς και να διαπραγματευτεί ένα νέο, μια νέα συμφωνία ΠΟΕ για τα περιβαλλοντικά αγαθά. Η πρόσβαση της Κίνας στην νέα Διεθνή Συμφωνία για τις Κυβερνητικές Προμήθειες είναι επίσης κάτι θετικό γιατί νομίζω ότι είμαστε οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και πρέπει να αποφεύγουμε τη λήψη προστατευτικών μέτρων. Να προσέχουμε να μην εφαρμόζονται τέτοιες, τέτοια μέτρα έτσι ώστε να συμβάλλουμε από κοινού στη δημιουργία ενός δίκαιου ανοιχτού παγκόσμιου εμπορικού συστήματος. Πριν καταλήξω θα ήθελα να σας πω σύντομα και κάτι σημαντικό που το ξέρετε όμως. Ελπίζουμε η Ένωση να πάρει την απόφαση να χορηγήσει στην Κίνα το καθεστώς οικονομίας της αγοράς. Αναγνωρίζοντας δε το δυναμισμό, τη στρατηγική σημασία και τη συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, θέλουμε τώρα βλέπουμε τώρα νέο ενδιαφέρον και από την Κίνα και από την Ένωση για την προώθηση των κοινών συλλογικών μας συμφερόντων για την ενδυνάμωση της εταιρική μας σχέσης, της ειρήνης, της ανάπτυξης των μεταρρυθμίσεων και του παλιτισμού. Και προσβλέπουμε σε ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία με την ίντα και όλων ημών με ύψιλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρέσβη. Έχουμε οκτώ μιλητέ των κατάλαβων των mm. ομιλητών. Τρία λεπτά για καθέναν. Ο κύριο Βίγκλερ, ο οποίο είναι συγητής μα θα πάρει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την κυρία Πρέσβη που βρίσκεται εδώ μαζί μα σήμερα και που μα παρουσιάζει ποιες είναι οι απόψεις σα. Πολύ καλή η νέα εικόνα και πιστεύω ότι ισχύουν αυτά που είπατε για το New Normal, αυτό το νέο κανονικό πρότυπο, το νέο σημείο αναφοράς ε, στην ε, Κίνα. Τρεις ερωτήσεις θα ήθελα να σας απευθύνω από πλευρά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας για τη συνεργασία με την Κίνα και από τις εμπειρίες ε, που μας έχουν αναφέρει τα ευρωπαϊκά επιμέλητρια στην Κίνα και από τις, ενώσεις, ε, τις βιομηχανικές ενώσεις. Εξοχότητα αναφέρατε καταρχάς τις συμφωνίες επενδυτικών ε, συμφωνιών μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα σημαντικά λοιπόν θέματα που είναι επιτάπητος είναι το θέμα της βελτιωμένης πρόσβασης στην αγορά για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στην Κίνα. Έχουμε στο Κοινοβούλιο και στην Διεθνή Επιτροπή ε, Εμπορίου ε, αναφορές που λένε ότι οι, οι αλλοδοπές εταιρείε έχουν ακόμα εμπόδια, αντιμετωπίζουν εμπόδια και μάλιστα αντιμετωπίζουν και νέα εμπόδια σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητά τους στην Κίνα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να σημειωθεί πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή. Ποια είναι λοιπόν η απόψή σας εξοχότητα. Θα υπάρξει πρόοδος ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά, σε ό,τι αφορά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Δεύτερη ερώτηση, η οποία είναι αλληλένδετη και με την πρώτη, αλλά λίγο πιο στοχευμένη. Μιλήσατε για τις μεταρρυθμίσεις. Ένα σημαντικό τομέα ε, όπου γίνονται στην Κίνα σημαντικές και εντυπωσιακέ ε, μεταρρυθμίσεις είναι ο τραπεζικός κλάδος. Φυσικά όταν μιλάμε για τον τραπεζικό κλάδο δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε και για την τεχνολογία IT της κοινωνίας ε, των πληροφοριών που συνδέονται με την τεχνολογία. Και πρώτα απ' όλα στον τραπεζικό τομέα που είναι κρίσιμη σημασία. Κάποιες αναφορές αναφέρουν ε, ενδείξεις κλεισίματος της αγοράς IT IT για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ε, καταρχάς στον τομέα και στον κλάδο του IT. Έχετε να σχολιάσετε, έχετε πληροφορίες να μας δώσετε. Και τρίτον, εν συντομία, ξέρω ότι διεξαγάγεται στην Κίνα αυτή τη στιγμή μια σημαντική μεταρρύθμιση του υγειονομικού κλάδου, που είναι πάρα πολύ σημαντική λόγω του μεγέθους του κλάδου. Ένα σημαντικός ε, κλάδος είναι η φαρμακοβιομηχανίας και οι δυνατότητες που θα είχαν οι ευρωπαϊκές φάρμακα βιομηχανίες να συνεργαστούν στην ε, μεταρρύθμιση του υγειονομικού κλάδου στην Κίνα. Σας ευχαριστώ και πάλι σας συγχαίρω για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Σιγητά, ευχαριστούμε. Και τώρα η Σκιώδης. Η κυρία Μόσκα. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την πρέσβυρα για αυτή την ε, πλήρη απεικόνηση της οικονομικής κατάστασης και των ε, μεταρρυθμίσεων ε, που υλοποιεί η Κίνα. Εγώ έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την είδηση που όλοι διαβάσαμε πρόσφατα σε σχέση με την ε, Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων στο υποδομές με την προσχώρηση για κάποιων ευρωπαϊκών κρατών. Θα ήθελα κάποια περαιτέρω στοιχεία από την πρέσβυρα για το πώς αυτή η πρωτοβουλία μπαίνει στο πλαίσιο της ευρύτερης οικονομικής και γεωπολιτικής στρατηγικής που μας παρουσιάστηκε σήμερα. Μία δεύτερη ερώτηση αφορά ένα ζήτημα που έχουμε συζητήσει ευρέως ε, σήμερα το πρωί στην Επιτροπή μας, δηλαδή η αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων επειδή δεν ε, λάβαμε περαιτέρω ειδήσει μετά από το γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα από τον περασμένο Ιούνιο σε σχέση με τα βήματα που θα μπορούσαν ε, να γίνουν για το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν είμαστε σε μια κατάσταση τέλματος ή αν θα μπορούσαμε να αναμένουμε κάποιες προόδους ε, στην αμοιβή αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων και να δούμε και ποια είναι τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν και πρέπει να υπερβληθούν για την αμοιβαία αναγνώριση στο θέμα αυτό και πιο γενικά για το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Εμείς ως ευρωπαϊκή Ένωση κινούμαστε πολύ σε αυτό το θέμα και θα θέλαμε να ξέρουμε πώς και στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να βρούμε μια δυνατότητα συνεργασίας και μηδέας αναγνώρισης. Και μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με ένα σημείο που θέσατε, δηλαδή την αναγκαιότητα να μην έχουμε θέσεις προστατευτισμού, όπως αναφέρατε. Θα ήθελα μία διευκρίνηση για το ποια είναι η πρόθεσή σας. Το Φεβρουάριο του 2015 εντός του μηχανισμού του ΠΟΕ υπήρξε μία διακήρυξη επιβολής ε, δασμών ε, για τους σωλήνες χάλιβα. Θα ήθελα να μου πείτε από την πλευρά της Κίνας ε, Ποια είναι η πρόθεσή της, δηλαδή πρόκειται να άρει αυτούς ε, τους δασμούς που έχουν κριθεί ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ή θα πρέπει να κάνουμε έφεση εντός της προθεσμίας. Ευχαριστώ κύριε Σόλτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την κυρία Πρέσβη για την εκτενέστατη και στοχευμένη παρουσίαση της σημερινής ε, εμπορικής σχέσης και σχέσης συνεργασίας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω ότι όλοι ε, προσβλέπουμε στην εμβάνθυνση των ε, εμπορικών σχέσεων και είναι προς το συμφέρον όλων μας ε, όταν εκείνη λαμβάνει αποφάσεις τέτοιου είδους επηρεάζουν ασφαλώς έχουν αντικτύπωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν Προσβλέπω και στις δύο σημαντικές εκδηλώσεις ε, στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας και στο Εμπορικό Συμβούλιο Διαπραγματεύσεων στο φετινό έτος. Δύο ερωτήσεις λοιπόν θα είχα να απευθύνω προς την κυρία Πρέσβη. Σε ό,τι αφορά την επενδυτική συμφωνία με πρόσβαση στην αγορά όταν μιλάμε για θέματα της Αγιατικής Τράπεζας επενδύσεων και ανάπτυξης, όταν μιλάμε για θέματα υπέρβασης των δυσκολιών στις διμερείς σχέσεις. Πάντα μιλάμε ουσιαστικά για τον ε, ρεαλιστικό αντίκτυπο στην πράξη στις δύο χώρες. Για παράδειγμα, τα εργασιακά πρότυπα, πώς διαμορφώνονται. Η πολιτική απασχόληση, η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο μεγάλων αυτών ε, εμπορικών εταίρων, πώς διαμορφώνονται τα περιβαλλοντικά πρότυπα, πώς θα πρέπει να αναπτυχθούν στο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει όλη την κοινωνική ανάπτυξη και της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω, επειδή μιλήσατε για τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα, τι περιμένετε από τους επόμενους ε, διαπραγματευτικούς γύρους και από τις επενδυτικές συμφωνίες σε ό,τι αφορά και τις συγκεκριμένες ε, υποχρεώσεις των ε, επενδυτών που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη θητεία για να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Και επίσης ε, για την ενίσχυση των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του ΠΟΕ και σε ό,τι αφορά τους γύρους της Δόχα. Στο άμεσο μέλλον θα ήθελα να ξέρω πού πιστεύετε ότι μπορούν να υπάρξουν συγκεκριμένα σημεία αναφοράς και σε ό,τι αφορά το υπουργικό, την υπουργική συνάντηση, την υπουργική σύνοδο στα τέλη του έτου στην Κένια. Πού πιστεύετε λοιπόν ότι εστιάζονται τα προβλήματα της διεθνούς οικονομίας και πού μπορούν η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας και η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού να βοηθήσουν στην υπερβασόν εμποδία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπούχνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρέσβη. Αναφερθήκατε στην προστασία των επενδύσεων. Όπως ξέρετε ασκείται μεγάλη κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ISTS. Και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να μεταρρυθμίσει το εργαλείο αυτό. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει και θα θα πρέπει άμεσα να βελτιωθεί. Δεύτερο θέμα, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα θέμα μη διαπραγματεύσιο για την ομάδα μου αλλά και για όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χωρίς μια δέσμευση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το Κοινοβούλιο να συμφωνήσει και να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Συνήθως οι πράσινοι θεωρούν ότι η συμπληρωματική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπερβολικά αδύναμη γιατί δεν περιλαμβάνει ένα μηχανισμό εφαρμογής των δεσμεύσεων από πλευρά των συμβαλόμενων μερών. Για μας ε, ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών, ε, αστικών διαφορών είναι ένα θέμα που αποτελεί κόκκινη γραμμή σε ό,τι αφορά περίπτωσης ε, σοβαρών παραβιάσεων, η κυβέρνηση σας πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αναλάβει τέτοιες δεσμεύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Ντάρτμουθ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν, πρέπει να συγχαρώ την πρέσβυρα για την γλαφυρότητά της ε, και μπορώ να πω ότι ε, πολύ καλύτερη τα προφάτησα από τη δική μου και δίκιο είχε αποδώσει έμφαση στο εμπόριο γιατί έχουμε μεγάλο όγκο εμπορίου μεταξύ της ε, Κίνας και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε πάνω από ένα δισεκατομμύριο την ημέρα. Εγώ, εγώ έχω 428 δισεκατομμύρια το 2013 και στις εξαγωγές έχουμε 220 ε, δις. Μεγάλος όγκος λοιπόν. Και αυτό ε, ε, κάποιοι στη χώρα μου ε, πώς θα έβλεπαν ε, ότι θα γινόταν αυτό το εμπόριο χωρίς δεν ήμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλοί εξαπατούν τους ψηφοφόρους λέγοντας ότι πρέπει να ε, είσαι μέλος ε, μια πολιτικής Ένωση για να μπορείς να κάνεις εμπόριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών, όπως είπε και η πρέσβυρα, η Νέα έχει μια τέτοια συμφωνία με την Κίνα και η Αυστραλία. Ακόμα και η Ισλανδία έχει συμφωνία ελεύθερο εμπορίου με την Κίνα, αλλά αυτός που δεν έχει συμφωνία ε, ελεύθερου εμπορίου είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, δεν είναι και πολύ πιθανό να γίνει μια τέτοια συμφωνία. Αναφέρθηκε από κάποιο προλελήσατε. Τώρα έχω μια ερώτηση για την πρέσβυρα. Στο παρελθόν μιλήσαμε για ε, την ε, επιβολή του νόμου σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία σε τρίτε χώρε. Ε, και έχω κάποιου εκπροσωπού από τη μουσική βιομηχανία που ανησυχούν πάρα πολύ ε, για το πώ η διανοητική ιδιοκτησία ε, παραβιάζεται συνεχώς στην Κίνα, στον τομέα της μουσικής και μπορώ να πω υπάρχει κάποια λογική προοπτική η κυβέρνηση της Κίνας να τηρήσει και να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ας μιλήσουμε απλώ για τη μουσική. Ας μην μιλήσουμε τώρα για τα φάρμακα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σίκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Λεκρός Τσίκου. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος ε, από τα όσα θέλησε να προτείνει η πρέσβυρα στην Επιτροπή μας και εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι η Κίνα σίγουρα αποτελεί μια αγορά η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική και πολύ μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης και ελκύει τους Ευρωπαίους επενδυτές. Έχουν γίνει κάποια βήματα προς τα μπρος και φυσικά είναι ιδιαίτερα σκόπιμα. Και επομένως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς θα δώσουμε μια προοπτική σε αυτά τα βήματα πρόοδου. Θέλω και εγώ λοιπόν να κάνω κάποιες ερωτήσεις ε, προς την πρέσβυρα, αλλά και κάποιες συστάσεις. Γιατί εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει και να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται για να εγγυθούμε μια σωστή εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ, κυρίως σε ό,τι αφορά την απαγόρευση των κρατικών επιχορηγήσεων στις εξαγωγές και ε, την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διανοητική διοκτήσια Και επίσης, ε, τι γίνεται ε, προκειμένου να μπορούν όλοι οι εμπορικοί εταίροι να χαίρουν των ίδιων συνθήκων μεταχείρισης σε ό,τι αφορά και την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Για να ανοίξει η αγορά σε ξένες υπηρεσίες και εμπορεύματα ίσως χρειάζονται πιο μεγάλες και διαφανείς εγγύησεις ε, από το θέμα της συμμετοχής ε, στις δημόσιες προμήθειες και των αλλοδαπών εταιριών. Και επίσης έχουν γίνει πολλά βήματα από την Κίνα για την προστασία του περιβάλλοντος και προς τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς προβλέπετε βέβαια σε αυτή την περιβαλλοντική πτυχή. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Ροντρίγες. Ευχαριστούμε την πρέσβυρα που είναι εδώ μαζί μας. Θα ήθελα να Κάνω τέσσερις ερωτήσει συγκεκριμένε. Καταρχήν, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψη και το όραμα που έχει η πρέσβυρα της Κίνας σε σχέση με το πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε πράγματι στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Φυσικά ε, ξεκινώντας έχοντας ε, ως εφετηρία πολύ διαφορετικές ε, συνθήκες σε ό,τι αφορά τους κανόνες και τα πρότυπα που πρέπει να σεβαστούν και δύο πλευρές. Η δεύτερη ερώτηση. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω αν μπορείτε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για το ποιο είναι το σημερινό στάδιο των διαπραγματεύσεων και τι γεωγραφικέ ενδείξει. Τρίτον, σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις. Όποια οικονομία θέλει να είναι οικονομία της αγοράς, φυσικά πρέπει να ανοίξει και τον κλάδο των δημοσίων συμβάσεων. Θα ήθελα λοιπόν πράγματι να ξέρω σε ποιο σημείο οι διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά θα οδηγηθούν από την πλευρά της Κίνας ε, και ε, πράγματι θα πρέπει να γίνει απελευθέρωση των θεωρήσεων έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε project και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην Κίνα. Ναι. Σε σχέση με το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς, θα ήθελα να ξέρω μέχρι ποιο σημείο έχει προωθήσει η Κίνα την πολιτική ε, καθορισμού τιμών σε σχέση με τις συνθήκες ελεύθερης προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών και ζήτησης. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Αν επιτρέπετε, κυρία Πρέσβη, θα ήθελα και εγώ να σας θέσω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση σε ό,τι αφορά το καθεστώς οικονομίας της αγοράς. Πέντε κριτήρια προβλέπονται, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται. Η Κίνα μπορεί να αποδείξει ότι τα πέντε αυτά κριτήρια όντως πληρούνται γιατί αυτά αποτελούν ε, το βασικό, τη βασική προϋπόθεση προκειμένου να χορηγηθεί το καθεστώς οικονομίας αγοράς. Δεύτερη ερώτηση. Με τη συμφωνία στον Παλή και με τις σαφείς συζητήσει για τις διευκολύνσεις στο εμπόριο, υπήρξε κάποια μικρή κίνηση στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ. Ποια πιστεύετε ότι είναι η θέση και ο ρόλος ε, της Κίνας εν ώψη και της Υπουργικής Συνόδου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της εμπορικής διευκόλυνσης και σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες ε, μελλοντικές συμφωνίες στα πλαίσια του ΠΟΕ. Τρίτη ερώτηση. Παρατηρείτε πιο πολύ αύξηση μάλλον των άμεσων ε, κινέζικων επενδύσεων στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν, επενδύσει δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να ακούσω από πλευρά σας πώς αξιολογείτε τις επενδυτικέ δυνατότητες και τις, ε, τους όρους, ε, τα θέματα νομικής βεβαιότητας και ασφάλειας ε, στην Ευρώπη προκειμένου να προσελκύσουμε κινέζικες επενδύσεις ε, στην Ευρώπη. Και τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Μπέτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Πρέσβη για την πολύ καλή παρουσίαση. Από δική μα πλευρά θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι ε, είναι εντατικό το ότι η δεσμευσή μα με την Κίνα σε όλα τα επίπεδα, διμερό, πολυμερό. Η Κίνα είναι σχεδόν ο μεγαλύτερο εταίρο, ο εμπορικό εταίριο. Ένα δισεκατομμύρια ε, ευρώ ανά ημέρα, λέμε συνήθω. Εστιαζόμαστε σε αυτό, αλλά υπάρχει πολύ μεγαλύτερο δυναμικό σε ό,τι αφορά την εξίσωση των όρων πρόσβασης στην αγορά. Σε ό,τι αφορά την επενδυτική πλευρά, το κάνουμε μέσω διμερών συμφωνιών. Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίε, το κάνουμε επίσης και σε ό,τι αφορά τις, ε, την ανάθεση συμβάσεων. Με την σχετική συμφωνία για τις ε, συμβάσεις μέσω ε, πολυμερών ε, σχέσεων το κάνουμε αυτό για τους ε, δασμολογικούς φραγμούς και σε ό,τι αφορά την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων μέσω του διαλόγου IP στο 10ο πλέον έτος και μέσω των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για τη γεωγραφική προέλευση όπου έχουμε ακόμα πολλές, πολλούς όρους να αντιμετωπίσουμε. Καλωσορίζουμε όντως ε, την πρόοδο που σημειώνεται στην Κίνα από τον Πρόεδρο. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις ε, στην Κίνα, τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει και ο κόσμος και ο λαός, αλλά και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό θα πάρει χρόνο. Κοιτώντας ε, με χρονικό ορίζοντα το 2020, ξέρουμε ότι αυτά θα πάρουν χρόνο, αλλά ελπίζουμε ότι η εμβάθυνση των εμπορικών μας ε, σχέσεων με την Κίνα και το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς θα αλληλοϊποστρίξουν τα συμφέροντά μας προκειμένου να είναι εποφελής στη σχέση. Η ατζέντα μας είναι σαφή σε ό,τι αφορά το 2013 δημιουργήσαμε την ατζέντα 2020. Βασικό εμπορικό στοιχείο είναι η σύναψη και η ολοκλήρωση του πέμπτου γύρου των εμπορικών ε, διαπραγματεύσεων. Είχαμε ένα πολύ επικοδομητικό διάλογο. Τώρα προσβλέπουμε στον έκτο γύρο. Ελπίζουμε να έχουμε το σχετικό κείμενο και ε, στα τέλη του έτους να κάνουμε και τις συζητήσεις για την πρόσβαση στην αγορά. Στα τέλη του Ιουνίου, όπως αναφέρθηκε, θα γίνει η Σύνδοση Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα εδώ στις Βρυξέλλες και ο υψηλού επίπεδου οικονομικός και εμπορικός διάλογος στο Πεκίνο μετά το καλοκαίρι. Προσβλέπουμε στη συνέχιση των εργασιών μας για την ευάθυνση των εμπορικών μας σχέσεων με την Κίνα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα... Η κυρία Πρέσβης. You have another... Έχετε άλλα 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές. Όλες αυτές τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι είναι αδύνατη η αποστολή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Πολλές από τις ερωτήσεις που τέθηκαν σχετίζονται με αυτή την ε, σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Όπως είπα, αυτό είναι ένα εγχείρημα που θα είναι προς το συμφέρον και το δυο μας. Ε, εν τέλει δηλαδή θα είναι ένα θετικό σενάριο για όλους και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Εγώ προσωπικά δεν ε, έχω συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, δεν γνωρίζω πολύ καλά τις λεπτομέρειες. Απλώς μπορώ να πω ότι είμαι επιπισμένη για την επιτυχή έκβαση αυτής της Σφαιρικής Συμφωνίας Επενδύσεων. Γιατί, όπως είπα, αυτό εξυπηρετεί τα θεμελιώδη συμφέροντά μας. Και θα είναι μια σφαιρική συμφωνία επενδύσεων. Νομίζω ότι κάποια από τα θέματα που τέθηκαν στις ερωτήσεις θα καλυφθούν. Ο σκοπός είναι να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη πρόσβαση και στις διαγορές και της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρασχεθεί ισχυρή προστασία στους επενδυτές δυνάμει της συμφωνίας. Όπως ε, είπε και ο συνάδελφος μόλις τώρα, οι διαπραγματεύσεις αυτές προδεύουν καλά και όλοι όσοι συμμετέχουν έχουν δεσμευτεί πλήρως για να συνεργαστούν προκειμένου να υπάρχει μια επιτυχής έκβαση. Υπήρχε μια ερώτηση για την ασιατική ε, τράπεζα επενδυτικών υποδομών. Αυτή η τράπεζα δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες, ε, κυρίως στην Ασία, για ε, διασυνδεσιμότητα των υποδομών. Γιατί στην Ασία έχουμε ανάπτυξη, είναι μια δυναμική περιοχή και υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για επενδύσει σε υποδομέ. Δεν υπάρχει έλλειψη πόρων, αλλά υπάρχει έλλειψη ενός συστήματος χρηματοδότησης. Και η χρηματοδότηση από τους εφιστάμενους ε, χρηματοδοτικούς φορείς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν ε, επαρκούν για μια τέτοια ανάγκη. Αυτό λοιπόν θα ωφελήσει την περιφέρεια. Και αυτή η τράπεζα είναι μια ανοιχτή, διαφανής τράπεζα αναπτυξιακή. Θα επικεντρωθεί στις επενδύσεις σε υποδομές στην Ασία κυρίως και θα προωθήσει την περιφερειακή διασυνθησιμότητα και την οικονομική ολοκλήρωση. Mm. Από όσο γνωρίζω μέχρι τώρα, υπάρχουν περίπου 46 ή 47 ιδρυτικά μέλη. Υποθέτω ότι εργάζονται επί της χάρτας, επί του μηχανισμού λήψης αποφάσεων, επί ε, της ε, κατανομής, επιμερισμένης κατανομής. Αλλά οι αποφάσεις ε, θα λαμβάνονται ομόφωνα και θα γίνει αυτή μια τράπεζα διεθνούς προτύπου που θα χαρακτηρίζεται από το clean, από καθαρό και πράσινο επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα. Και επίσης ε, έχουμε κάποιες εμπειρίες ε, όπως το χάρη την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, την ε, Επενδυτική Τράπεζα στην Ασία. Έτσι λοιπόν αυτή η νέα τράπεζα θα βελτιώσει το συντονισμό με του υφιστάμενους πολυμερείς οργανισμούς και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε αμοιβαίο όφελος για όλους και δεν θα υπάρχει αποκλεισμό. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ για αυτή την επενδυτική τράπεζα. Και υπήρχε και μια ερώτηση σε σχέση με τη φορά το άνοιγμα της Κίνας. Αν διαβάσετε την ομιλία ε, πριν από ένα μήνα που εκφώνησε ο Πρωθυπουργό, η Κίνα θα προβεί σε ένα νέο άνοιγμα υψηλή ποιότητα. Πιο γρήγορα θα κινηθούμε προς να οικοδομήσουμε μια νέα ανοιχτή οικονομία. Μόλις ε, ανέφερα ότι ε, θα μεταμορφώσουμε το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας ε, και θα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς θα χρησιμοποιούμε το ξένο κεφάλαιο και πώς θα καταστήσουμε τους τομείς των υπηρεσιών και τις μεταποίησης πιο ανοιχτούς. Υπάρχει τώρα νομίζω μία αποστολή ε, του Κοινοβουλίου για το θέμα της υγείας. Θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στις ε, υπηρεσίες. Και όπως σας είπα θέλουμε λοιπόν να ανοίξουμε περισσότερο τον τομέα των υπηρεσιών. Επίσης θα εισαγάγουμε ένα σύστημα διαχείρισης για τα επενδυτικά έργα. Η Κίνα σίγουρα έχει ευνοηθεί πάρα πολύ από το άνοιγμα και αυτή την οδό θα ακολουθήσουμε, οπότε δεν θα κλείσουμε την πόρτα μας, θα την κρατήσουμε ακόμη πιο ανοιχτή. Και υπήρχε και μια ερώτηση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Εκφράστηκαν πολλές ανησυχίες για την επάρκεια της προστασίας των διανοητικών δικαιωμάτων στην Κίνα. Η απάντησή μου είναι, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα πιστεύει, ότι η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι ζωτικές για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και είναι πολύ σημαντικό να προστατευθούν ε, ε, αυτά τα δύο προς το συμφέρον της οικονομικής ανάπτυξης. Και φυσικά και η Κίνα έχει κάποια προβλήματα, όπως και άλλες χώρες, σε σχέση με την προστασία των γεωματών βηματικής διοκτησίας. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και κατά νου τις μεγάλες προσπάθειες που έχει καταβάλει η κυβέρνηση της Κίνας και τα μεγάλα επιτεύγματα τα οποία σημειώσαμε τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι στο χέρι μας για να προστατεύουμε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει και μια ανησυχία. Σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα και τον κλάδο της τεχνολογίας των πληροφοριών. Δεν κατάλαβα πολύ καλά την ερώτηση αυτή, αλλά θα σας πω κάποια πράγματα. Καταρχήν η Κίνα έχει δεσμευτεί στο άνοιγμα, όπως σας είπα, και το διαδίκτυο της Κίνας είναι ανοιχτό. Επομένως έχουμε μία αγορά διαδικτύου. Έχουμε χρησιμοποιήσει ευρέως τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στην Κίνα. Και επίσης φυσικά μας απασχολεί και το θέμα της ασφάλειας στον χώρο. Γιατί αυτή είναι μια κοινή παγκόσμια πρόκληση και για την Κίνα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετωπίζουμε και την πρόκληση της ε, ασφάλειας στο διαδίκτυο. Συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες σε αυτό. Η Κίνα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών του ίντερνετ. Περίπου 400 εκατομμύρια. Επίσης, είμαστε ταυτόχρονα και θύμα κυβερνοεπιθέσεων και έχουμε και καθυστερήσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών διαδικτύου. Θα πρέπει να εξορροπήσουμε την ανάγκη του να αναπτύξουμε τεχνολογίες ε, πληροφοριών και να προστατεύσουμε και την ασφάλεια του διαδικτύου. Έχουμε λάβει μέτρα όπως παραδείγματο χάρη κατάρτιση εθνικών στρατηγικών νόμων, κανονισμών που να αναπτύξουμε τεχνολογίες, IT και κυβερνοασφάλειας καθώς και να προωθήσουμε τις ε, ικανότητες για να χρησιμοποιήσουμε ε, και να διευρύνουμε τη διάδοση των πληροφοριών. Νομίζω το ίδιο κάνετε και εδώ στην Ευρώπη. Και τέλος η Κίνα θα προστατεύσει τα ένομα συμφέροντα των πολιτών τη και τα ενώμα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον νόμο. Και καλωσορίζουμε και υποστηρίζουμε τις ξένες εταιρείες και τις εταιρείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έλθουν στην Κίνα και να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους. Υπήρχε και μία ερώτηση για την προστασία του περιβάλλοντος Αν διαβάσετε τα στοιχεία θα δείτε τα μεγάλα επιτεύγματα της Κίνας. Πέρσι περιορίσαμε το διοξίδιο του άνθρακα, την ένταση του διοξίδιου του άνθρακα, πάνω από 3% και μειώσαμε ε, και τις ε, εκπομπές κατά 2% νητροδών και αμμονίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να μαχόμαστε κατά της ρήπανσης της ατμόσφαιρας και θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Επίσης, ε, θα ε, διευρύνουμε την δυνατότητα εμπορίας εκπομπών και θα ε, χρησιμοποιήσουμε και ενέργεια που να προέρχεται από βιομάζα, η αιωλική ενέργεια. Επίσης θα εκμεταλλευτούμε το σχιστολιθικό αέριο και θα συνεχίσουμε να βάλουμε το όριο στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και θα προωθήσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας στη μεταποίηση, στις μεταφορές και στην οικοδομή. Υπήρξε και άλλη μία ερώτηση σε σχέση με την διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι επί του οποίου εργαζόμαστε. Πριν λίγες μέρες είχαμε τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πεκίνο. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε εσωτερικό επίπεδο πρέπει να προβεί σε συντονισμό, γιατί τώρα είναι 28 τα κράτη-μέλη και αυτό χρειάζεται χρόνο. Όμως νομίζω ότι σημαίνουμε πολύ καλή πρόοδο και ελπίζω ότι πριν την επόμενη Σύνοδο μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουμε μπορέσει να σημειώσουμε πραγματική πρόοδο στο θέμα της διευκόλυνσης ε, χορήγησης θεωρήσεων. γιατί φυσικά αυτό θα διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές μας. Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις θα καλέσω τους αδέλφους να πάρουν το λόγο. Α, συγγνώμη, για τη γεωγραφική ένδειξη, μάλιστα. Η Κίνα είναι αρκετά ικανοποιημένη με τη σημερινή διαδικασία διμερών διαπραγματεύσεων για την ε, σύναψη συμφωνία συνεργασία για το θέμα αυτό και τα δύο μέρη μέσω των διαπραγματεύσεων ε, έχουν επισημάνει κάποια τεχνικά προβλήματα. Έχουμε εντοπίσει τομεί σημαντικού για τη μελλοντική δουλειά. Ελπίζει η Κίνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να δείξει ευελιξία για να επιληθούν τα εκκρεμή ζητήματα θα θέλαμε να συνεχίσουμε το διάλογο και την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν επικοδομητικό και ρεαλιστικό τρόπο και να προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να έχουμε αμοιβαία ωφέλιμα αποτελέσματα. Η Κίνα για την επίλυση διαφορών κράτους επενδυτή πιστεύει ότι αυτό θα προστατεύσει θετικά τα συμφέροντα των επενδυτών και το θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική συνιστόσα στο διεθνές σύστημα. Εδώ και δεκάδες χρόνια η πρακτική μας έχει δείξει ότι το σημερινό σύστημα ESDS έχει ελαττώματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν επιγόντως. Ελπίζει λοιπόν η Κίνα ότι θα μπορέσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μηχανισμό επίλυσης διαφορών που θα είναι λειτουργικός. Θα πρέπει λοιπόν να καινοτομήσουμε για το SDS. Okay. And with regard to the uh, σε ό,τι αφορά τώρα το καθεστώς ε, οικονομίας αγοράς, αυτό δεν είναι κάτι διμερές. Είναι κάτι που γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Η Κίνα θα αποκτήσει αυτό το καθεστώς οικονομίας της αγοράς το 2016, του χρόνου, σύμφωνα με τον ΠΟΕ. Ελπίζουμε λοιπόν ότι και οι δύο πλευρές θα σεβαστούν τους κανόνες του ΠΟΕ και θα καταπολεμήσουν τον προστατευτισμό και δεν θα χρησιμοποιήσουν αμυντικά εμπορικά μέσα. Εγώ πιστεύω ότι η Κίνα έχει σεβαστεί όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει ένα έθνος ε, οικονομίας της αγοράς. Ορισμένα από τα κριτήρια έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή σας θα διδραματίσει θετικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. για να ληφθεί μια επίσημη υπόφαση για να χορηγηθεί στην Κίνα αυτό το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς. Okay. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πρέσβη. Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά που σας είχαμε εδώ κοντά μας. Και τώρα το λόγο έχει ο κ. Βέγκλερ, ο οποίος είναι μόνιμος σε Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εξοχότητη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο, παρά μόνο να εκφράσω την ειλικρινή επιθυμία της Επιτροπής μας να συνεργαστούμε μαζί σας, προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος ε, τις διαπραγματεύσεις ε, που διεξαγάγονται. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο έχει νέες εξουσίες ε, βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά πάντα τονίζουμε ότι και η εξουσία εποπτείας των περιστατικών συμμετοχής διαπραγματεύσεων και διατύπωσης μιας τοποθέτησης αποτελεί νέα αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο θα ασκήσει τα δικαιώματά του αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Θα παραμείνουμε σε επαφή και θα τα πούμε σύντομα, πιστεύω. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Okay, now we are moving back to 16. Πάμε πάλι λοιπόν τώρα στο σημείο 16, στην ομάδα παρακολούθησης. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι ομάδες παρακολούθησης δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντικές ε, για να παρακολουθούμε τις ε, εξελίξεις, για παράδειγμα, την διαπραγματεύσεων με την Κίνα, και επειδή είναι λοιπόν τόσο σημαντικές αυτές οι ομάδες, θα πρέπει να συντονίζουμε τις εργασίες μας. Η σύσταση δε των ομάδων αυτών παρακολούθησης θα πρέπει να συνοδεύεται από ενημέρωση και συντονισμό. Είναι υποδειγματικό λοιπόν αυτό το μοντέλο και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την καλή συνήθεια. Μεξικό. 26 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα. Ο κ. Μόιζερ, ο εισηγητής μας, ήταν και στην αντιπροσωπεία με το Μεξικό. Please. Yes, Sorry, I was busy. Πρόεδρε, ναι, συγγνώμη, μιλούσα εδώ πέρα με τη συντονίστρια. Και τώρα μικροφωνίζω, μάλιστα. So, uh, we had a very good... Λοιπόν, οργανώθηκε μια πολύ καλή ομάδα επιτήρησης για το Μεξικό στις 26 Φεβρουαρίου λίγες μέρες μετά περιμένω να φύγουν ησύχως. Ησυχάστε παρακαλώ. Είπα θα είμαι σύντομος αλλά ελπίζω και ενδιαφέρον. Λοιπόν, είχε οργανωθεί επίτηδες μερικές μέρες μετά τη συνάντηση του Κοινής κοινοβουλευτική Επιτροπή Επιτροπής στο Μεξικό όπου είχα τη τιμή να εκπροσωπώ την Ίντα. Εξαιρετικό γεγονός αυτό για το Κοινοβούλιο να στείλει εκπρόσωπο της Ίντα στην μεικτή κοινοβουλευτική. Πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση για την περιγραφή της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης στο Μεξικό συγκρίσιμη αυτή τη στιγμή των διαπραγματεύσεων ή προδιαπραγματεύσεων για τον εξυγχρονισμό τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών που είναι τμήμα της φερική συμφωνία που έχουμε με το Μεξικό από το 2000. Επίση Επίσης έκανα μία διμερή συνάντηση στο Μεξικό με τον ε, Υφυπουργό Φραντσίσκο Ρόζενσβάικ που ασχολείται με το εξωτερικό εμπόριο στο Μεξικό. Είναι ο κύριος διαπραγματευτής και έδωσα στο Μεξικό ένα μήνυμα και στους κοινοβουλευτικούς και στη δημόσια διοίκηση εκ μέρους της Επιτρόπου Μάλφτρομ που ε, ήθελε να επιδείξει καθαρά την πολιτική θέληση να φτάσουμε στην αναθέρμανση των διαπραγματεύσεων ή μάλλον στην αρχή των διαπραγματεύσεων για τον εξυγχρονισμό της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών. Το πρώτο τμήμα της συνεδρίασης ήταν πληροφοριακό για αυτή τη μεικτή κοινοβουλευτική όπως σας είπα και μετά έγινε μια πολύ ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Κομισιών και του, υπουργού, του πρέσβη Χουάν Καμάτσο το... και τα κύρια στοιχεία θα σας τα πω σε λίγο. Τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που έθιξε ο πρεσβευτής ήταν τα εξής. Το εμπόριο με τον ναύτα είναι πια τμήμα του DNA του Μεξικού, του δεσοξυριβοζωνουκλεϊκού οξέως του Μεξικού. Και ιδιαίτερα οι σχέσεις του με την Ένωση υπό την κυβέρνηση Ανανιέτο έχουν γίνει τεράστιες μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς που ιστορικά πάντοτε προστατεύονταν, υπήρχαν μονοπόλια δηλαδή στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες και έτσι δημιουργήθηκαν τεράστιες ευκαιρίες για ε, αμερικανικές αλλά και ευρωπαϊκές εταιρείες. Σήμερα ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Μεξικού είναι η Κίνα και όχι πια η Ένωση, χάνουμε δηλαδή μερίδια της αγοράς καθώς το Μεξικό διαπραγματεύεται και άλλες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των οποίων και το TTIP. Έχει σχεδιάσει ένα τεράστιο πρόγραμμα υποδομών ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων αν θυμάμαι καλά πράγμα το οποίο βέβαια καθιστά το άνοιγμα της αγοράς δημοσίων προμηθειών για ευρωπαϊκές εταιρείες κάτι πολύ ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά το Μεξικό δεν είναι ικανοποιημένο με την αργή όπως λέει πρόοδο των διαπραγματεύσεων και των προτεραιοτήτων που, στους οποίες θα βασιστεί η διαπραγμάτευση. Απ' την άλλη η Κομισιόν σας είπα, ήταν πολύ ειλικρινής η ανταλλαγή απόψεων η Κομισιόν. Είπε και αυτή μερικά σημαντικά πράγματα. Επειδή η συμφωνία υπάρχει μεν αλλά εξυγχρονίζεται και βάσει αυτής οι αριθμοί των συναλλαγών μεταξύ Ένωσης και Μεξικού έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Για να έχει νόημα η αναδιαπραγμάτευση πρέπει να έχουμε φιλόδοξους στόχους. Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης δεν θα είναι γρήγορα, δεν θα έρθουν γρήγορα βέβαια, εκτός αν είμαστε πολύ φιλόδοξοι και καλύπτουμε πάρα πολλούς τομείς. Και το Μεξικό απαντάει ότι και τα μυντικά και τα επιθετικά συμφέροντα πρέπει να καλυφθούν. Η μια πλευρά μπορεί να θελήσει περισσότερα στοιχεία που να την συμφέρουν και το ίδιο θα κάνει και η άλλη. Αυτό είναι φυσικό. Συζητήσαμε επίσης την ανάγκη να δούμε τι διαφορές υπάρχουν εμπορικά μεταξύ μας. Δεν συνδέονται τόσο πολύ με τον εξυγχρονισμό της, την ενημέρωση της συμφωνίας, αλλά θέματα όπως την πρόσβαση της Κροατίας στην Σφαιρική Συμφωνία που θα οδηγήσει σε ορισμένες ζημίες για το Μεξικό, όχι όμως τεράστιες, από τους δασμούς. Τώρα και οι δύο πλευρές επέδειξαν σαφή θέληση και πολιτικός και τεχνικός να υπάρξει επιτάχυνση για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα μέχρι το καλοκαίρι. Και πράγματι μετά την συνεδρία της ομάδας αυτής που έγινε στις 26 Φεβρουαρίου έγινε και μια άλλη πλήρης ανταλλαγή απόψεων Μεξικού και Κομισιόν για την κοινή έκθεση. Οργανώνονται σύντομα και άλλες συναντήσεις και αυτή την εβδομάδα τεχνικές και πολιτικές για να προχωρήσουμε με την Joint Vision Report, με την έκθεση κοινού οράματος. έτσι ώστε να τελειώσουν όλα το καλοκαίρι. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι η διαδικασία προχωράει καλά, αλλά βέβαια θα δούμε. Πιστεύω ότι μέχρι να έρθει τον Ιούλιο ο πρόεδρος Πανανιέτο πράγμα το οποίο βέβαια μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι να έρθει λοιπόν τελεία. και είμαι πεπισμένο ότι η Κομισιόν θα κάνει ό,τι πρέπει για να υπάρξει κατάληξη μέχρι το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι η διαδικασία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και αν έχετε απορίες να σας τις λύσω με τα χαράς και για την κοινή κοινοβουλευτική και για τα άλλα θέματα. Ξέραμε ότι είναι σημαντικό το θέμα και το πρόβλημα, ή ο εξυγχρονισμός δηλαδή τη υπάρχουσας συμφωνίας. Τεχνικά είναι πολύ σημαντικό οι μόνιμοι εισηγητές μας να πηγαίνουν στην αντιπροσωπεία γιατί έχουν την απαραίτητη γνώση και έτσι μπορούν να κάνουν σαφείς και ρητές δηλώσεις. Πρέπει πάντοτε να πηγαίνουμε λοιπόν. Καναδάς. Η ομάδα επιτήρησης συνεδρίασε αρχές Μαρτίου με τον Φιλίπ Τζουπουή αρχιδιαπραγματευτή. Συζητήθηκαν θέματα προμηθειών IPR, κανόνων προέλευσης και ο εισηγητής μας εδώ Έπρεπε να μας τα πει αλλά λείπει. Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων έγινε επίσης μια συνεδρίαση στις 3 Μαρτίου. Ο κύριος Φιέλνερ έχει λεπτομέρειες γι' αυτό. Ηνωμένε Πολιτείε συνάντηση 21 Μαρτίου με την Μόνικα Χένσκι υπεύθυνη τμήματάρχηδα για την βιώσιμη ανάπτυξη και συζητήσαμε την, το, πιθανές κεφάλαιο, το πιθανό κεφάλαιο βιωσιμότητα στο TTIP. Η Ιαπωνία συνάντηση στις 21 Μαρτίου πάλι ο κύριος Πιέρα εδώ ε, Βέβαια Περέρα γνωρίζει περισσότερα, ορίστε. Να σας πω ότι είχαμε την ομάδα παρακολούθησης 24 Μαρτίου. Όπως το θυμάστε, ο ένατος γύριος διαπραγματεύσεων υλοποιήθηκε το Φεβρουάριο, αλλά ήδη είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε εδώ στην Επιτροπή και τον πρέσβη από την Ιαπωνία και τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό, επόμενος γύρος θα λάβει χώρα από τις 23 ως τις 28 Απριλίου. Σε αυτή την ομάδα παρακολούθησης είχαμε την ευκαιρία να ακούσαμε κάποιους, ε, κάποια μεγάλα ενδιαφερόμενα μέρη από την πλευρά της Ιαπωνίας. Ε, τώρα είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε την Ένωση Μεταποιητών της Ιαπωνίας και το ε, Επιχειρηματικό Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη από τους σιδηροδρόμους. Όλοι είχαν πολλά να πούν για τις διαπραγματεύσεις, ενδιαφέρονται πολύ για τη συμφωνία. Η Ιαπωνική Ένωση είπε ότι, μάλιστα ότι υποστηρίζει την ε, Ιαπωνική Συμφωνία Ελευθεροπορίου, ο κλάδος των σιδηροδρόμων είπε ότι η εταιρείε της Επινίας ε, ήδη ε, συμμετείχαν σε διαγωνισμούς ε, παγκοσμίω για την προμήθεια τροχαίου υλικού και επίσης σημείωσαν ότι η ρήτρα επιχειρησιακής ασφάλειας ήταν μια απόπειρα να επευληθούν κάποιες υπάρχουσες διαφορές. Επίσης, ε, η Ένωση των ε, κατασκευαστών αυτοκινήτων της αυτοβιομηχανίας ε, είπε ότι ήταν υπέρ του να συναυθεί γρήγορα μια συμφωνία Θεωρεί ότι αν βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον θα έχουν και καλύτερες δραστηριότητες. Επίσης έχουμε και το θέμα των key cars που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στις διαπραγματεύσεις αυτές που αφορούν την αυτοβιομηχανία. Έτσι λοιπόν, πολύ θετική ήταν η στάση των επάνω μερών. Απέναντι στις διαπραγματεύσεις φυσικά υπήρχαν διαφορές μεταξύ της προσέγγισης των Ευρωπαίων και των Ιαπώνων. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να αναφέρουμε ότι ε, ήταν ε, αργή η πρόδραση της διαπραγματεύσης τους τελευταίους μήνες. Ε, θα δούμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες και φυσικά και στη Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου τον επόμενο μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Ουκρανία. Είχαμε συνεδρίαση της Ομάδας Παρακολουθήσης 24 Μαρτίου με τον ε, αρμόδιο υπουργό της Ουκρανίας, τον υπουργό εμπορίου. Παρουσιάστηκαν προσπάθειες που γίνονται από την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Και γίνονται ε, ουσιαστικά ε, προσπάθειες για την επισφαιρική ξεβάθρωση συμφωνίας ελεύθερων Συνελλαγών. Συζητήθηκε και το θέμα των εμπορικών προτιμήσεων και της αποπληρωμής της μακροοικονομικής βοήθειας. Ο κ. Λασβέργκης είναι εισηγητής και θα μπορούσε να μας δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Κίνα. 25 Μαρτίου συναντήθηκε η ομάδα παρακολούθησης. Ο μόνιμος εισηγητής είναι εδώ δίπλα μου. Αγαπητέ συνάδελφοι, αγαπητέ Πρόεδρε. Ο κύριος Μόησερ νομίζω ότι έχει θέσει τα πρότυπα. Θα πρέπει να είμαστε και σύντομοι και ενδιαφέροντες. Δεν ξέρω αν θα με ενδιαφέρον, αλλά σίγουρα θα είμαι σύντομος. Γιατί. Μόλις έγινε ένας εκτενής διάλογος για την Κίνα και πολλά από τα στοιχεία τα οποία συζητήσαμε, συζητήθηκαν και στην ε, συνάντηση της ομάδας παρακολούθησης, η τρίτη της ε, ομάδας παρακολούθησης στην τρέχουσα θητεία. Όπως ε, και παλαιότερα έχουμε τον κύριο Γιώ Λάινεν, ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας με την Κίνα. Είχαμε και την εμπειρογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κύριο Σλέγκερμις, ο οποίος είναι ο κύριος διαπραγματευτής για την επενδυτική συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο εξέλιξεις συζητήσαμε. Η μία εξ αυτών είναι ο διάλογος εμπορικής συμφωνίας και εμπορίου με την Κίνα. Συζητήσαμε το θέμα του καθεστώτος οικονομίας αγοράς της Κίνας και φυσικά δεν ήταν σαφής η κατάσταση όπως μας την παρουσίασε η αξιότιμη πρέσβης της Κίνας γιατί το θέμα του καθεστώτος οικονομίας αγοράς από νομικής πλευράς είναι λίγο πιο περίπλοκο. Ενημερωθήκαμε επίσης ότι και οι υπηρεσίες ε, του Κοινοβουλίου αλλά και της Επιτροπής εξετάζουν το θέμα αυτό και ε, κατά πάσα πιθανότητα στο δεύτερο ήμιση του έτους θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα για το ποιο είναι το νομικό καθεστώς στην πραγματικότητα γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα είναι κάπως πιο περίπλοκα από αυτό που μας παρουσιάστηκαν πριν από λίγα λεπτά. Ένα δεύτερο θέμα είναι η συνολική επενδυτική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Είχαμε πέντε δύσκολους γύρους συζητήσεων. Επίκειται ο έκτος γύρος. Αν ε, ένα θέμα θα μπορούσα να αναφέρω, αυτό ήταν το θέμα του ISDS, της επίλυση διαφορών κράτους επενδυτού. Το έθιξε και η πρέσβης της Κίνας, η οποία κατανοεί ότι ένας μηχανισμός ε, προστασίας των επενδυτών θα πρέπει να αποτελεί τμήμα διμερούς συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία του μηχανισμού αυτού είναι υπό διαμόρφωση, να το θέσω έτσι. Αυτά λοιπόν, Πρόεδρε, αυτές είναι οι βασικές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα και σύντομος και συνεκτικός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το 16 της ημερήσιας διάταξης και τώρα λοιπόν να περάσουμε στο 18 ετήσια έκθεση για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Θα δώσω το λόγο παρά αυτά στον εισηγητή μας, τον κύριο Μπορέλη. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προφανές ότι η αρχή της επικορικότητας αποτελεί ένα από τους ακρογωνίους λίθους ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος στην βάση της ίδιας της ιδέας της Ευρώπης που περιλαμβάνεται στις συνθήκες και διέπει κάθε αρχή κοινή ανάπτυξης ε, συνδέεται και με την, το σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας λαμβάνει μια ε, νέα διάσταση αναζητώντας ε, μια δύσκολη ισορροπία μεταξύ όλων και περισσότερων αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκό επίπεδο και θέλουν οι πολίτε να έχουν περισσότερο έλεγχο επί των αποφάσεων που λαμβάνονται. Αυτό ε, μας οδηγεί στο πώς πρέπει να ερμηνεύουμε την αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα και με τα διδύματα που έρχονται από τα κάτω. Η αρχή της επικουρικότητας είναι οριζόντια σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην εμπορική πολιτική. Όμως αυτό που μπορεί να φαίνεται ως απλώς ένα παιχνίδι ευθύνης ουσιαστικά έχει μια συνιστότητα Ωστόσο, ουσιαστική που έχει αντίκτυπο σε όλου του πολίτες χωρίς μια σοβαρή ανάλυση του αντίκτυπου που ε, μπορούν να έχουν οι αποφάσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κινδυνεύουμε να απομακρύνουμε ακόμη περισσότερο τους πολίτες από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών ζητούν περισσότερη ενημέρωση και διάλογο με τα θεσμικά όργανα. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η πρόκληση της επικουρικότητας που αντιμετωπίζουμε σήμερα και με αυτό το πνεύμα συνειδητοποίηση θα σας παρουσιάσω ορισμένες σκέψεις που σχετίζονται με την έκθεση για την επικουρικότητα 2013. Θα επικεντρωθώ σε πέντε σημεία. Το πρώτο αφορά το ρόλο της επικουρικότητας στις, εμπορικές, στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βάσει των πολλαπλών συμφωνιών που συνάπτει με τρίτες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επικουρικότητα λαμβάνεται υπόψη συνήθως όταν υπάρχουν διατάξεις διεθνών συμφωνιών που έχουν αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο και απαιτούν από τα κράτη-μέλη να τοποθετηθούν. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε αποκλειστική ορμαδιότητα σε θέμα εμπορικής πολιτικής αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό ένα χώρο Αβεβαιότητα σε σχέση με διατάξεις που ε, αφαιρούν αποκλειστικά τι άμεσες ξένες επενδύσει, όπως έδειξαν διάφορες συμφωνίες με τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όπου μπορούν να υπάρχουν προβλήματα αρμοδιότητα, συγκρούσει αρμοδιότητας και υπάρχει λοιπόν αναγκαιότητα να το ξεκαθαρίσουμε ιδίω σε ορισμένου τομεί όπω τη ενέργεια. Ε, μία άλλη πτυχή αφορά τις ρήτρες διαφύλαξης και ε, το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή της επικουρικότητας. Το δεύτερο σημείο αφορά την ε, μακροοικονομική βοήθεια που είναι πλέον εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής Πολύ συχνά η ιδεολογική συζήτηση μας εμποδίζει να επικεντρωθούμε στα συγκεκριμένα αποτελέσματα και συνέπειες αυτής της βοήθειας. Το κριτήριο της αναλογικότητας μας ζητά να αξιολογήσουμε προσεκτικά αν οι προτάσεις μας μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμες για τους εταίρους που βοηθάμε. Φυσικά μετά από μια λεπτομερή εξάντη ανάλυση και κατόπιν έλεγχο του, του Κοινοβουλίου για τη χρήση ε, αυτών των ε, ε, πόρων. Μπορούμε να αναφέρουμε και την αρχή more for more που χρησιμοποιήθηκε απέναντι στο κράτη μετά την Αραβική Άνοιξη. Επίσης πρέπει να αναθεωρήσουμε τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η αξιολόγηση αντικτύπου, η μελέτη αντικτύπου εξάντε στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών. Πολλές φορές δυστυχώς έχουμε υπερβολικά αισιόδοξε μελέτες αντικτύπου και θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στην ε, TTIP. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν το 2013. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αξιολογήσουμε σε σχέση με αυτή την συμφωνία ποιος είναι ο αντίκτυπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ποιος θα ωφεληθεί πραγματικά. Μία συνθήκη, μία συμφωνία όπως η TTIP έχει φυσικά τεράστια πολιτική διάσταση, ε, αλλά είμαστε είμαστε σίγουροι ότι αυτή η συμφωνία είναι πράγματι χρήσιμη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχει θετικές συνέπειες για όλους εμάς και όχι μόνο για τις λίγες και μεγάλες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για το θέμα. Η απάντηση είναι όχι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γιατί οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν βάσει εκτιμήσεων που δεν μπορούν να αποδείξουν ούτε αποστικοποιήσουν σύμφωνα με τη μέθοδο ανάλυσης που ακολουθήθηκε από την Κομισιόν και επομένως εδώ η αρχή της επικουρικότητας της θα πρέπει να είναι στη βάση κάθε διαπραγμάτευση της Κομισιόν. Ένα άλλο σημείο που σχετίζεται με το προηγούμενο είναι αυτό του ISDS, επίλυση διαφορών κράτους επενδυτή. Εδώ ε, ουσιαστικά υπάρχει πάλι σύγκρουση συμφερόντων ε, μεταξύ ε, της εξουσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυριαρχίας των κρατών μιλών που ζητούν επιτακτικά να υπάρχει ανάλυση εις βάθος. Το τελευταίο σημείο με το οποίο θέλω να κλείσω έχει να κάνει με ένα θέμα που συνδέεται με την ίδια την καρδιά της επικουρικότητας. Είμαι πεπισμένο ότι ο καθένας από εμά εδώ στο Κοινοβούλιο δρά σύμφωνα με την εντολή που έχει λάβει από τους ψηφοφόρους να τους εκπροσωπήσει και να προστατεύσει τα συμφέροντά τους. Έτσι λοιπόν θέλω να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε το θέμα της επικουρικότητας κυρίως όταν μιλάμε για πολίτες και τοπικό επίπεδο. Θα ήθελα να επαναλάβω πόσο σημαντική είναι η εμπλοκή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε θέματα εμπορικά εμπορική πολιτική. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση τη επικουρικότητα. Οι πολίτε μα θέλουν να έχουν περισσότερε πληροφορίε και να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων κυρίως όταν υπάρχουν ε, ενδυνάμει συνάπειες ε, για τα άμεσα συμφέροντά τους. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά μέσα για να ε, συμμετέχουν οι πολίτες και για να του ενημερώσουμε. Έτσι, λοιπόν, δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε αυτό το στοιχείο. Δεν αρκεί το μέτρο της δημόσιας δεβούλευσης που χρησιμοποιεί η Κομισιόν. Είναι προφανές, γιατί δεν εγγυάται μια ισορροπημένη συμμετοχή. Αν οι αποφάσεις που λαμβάνουν τι Βρυξέλλες θέλουν να είναι τόσο πιο κοντά στους πολίτε σίγουρα θα είναι πιο αποτελεσματικές, αν είναι πιο κοντά θα είναι πιο αποτελεσματικές και συγκεκριμένες. Και εδώ ολοκληρώνω την έκθεσή μου και περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στους σκιώδες συζητητές ε, για δύο λεπτά στον καθένα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ ο Φερνάντο Ρούας, αλλά έχω την ομιλία του εδώ και θα τη διαβάσω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Βασιζόμαστε σε τρει κύριου στόχου. Πρώτον, να δούμε πώ οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα εφαρμόσουν αυτέ τι αρχέ Δεύτερον, να γίνει μια σύγκριση τη εφαρμοσιμότητα των προτάσεων με σύγκριση με προηγούμενε εκθέσει και τρίτον να γίνει μια ανάλυση των νομοδοτήσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων για τις προτάσει της Κομισιόν από το 2013. Από αυτή την άποψη η έκθεση θα έπρεπε να θεωρηθεί προσθήκη στην ετήσια έκθεση 13 της Κομισιόν για τη σχέση της με τα εθνικά κοινοβούλια. Με βάση την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που αναφέρει το άρθρο 5 of TFEU, we must... πρέπει να πούμε σε σχέση με το εμπόριο ότι οι αρχές αυτές έχουν κάποιο περιορισμούς λόγω των υπερβολικών δικαιοδοσιών που έχει η ενωσιακή εμπορική πολιτική. Η κυριότερη τομής που αφορά η συμφωνία είναι η αίτηση χρηματοπιστωτικής βοήθειας όταν και εφόσον υπάρξει βελτίωση εξάντε αξιολογήσεων ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αναλογικότητα και όπου η χρηματοπιστωτική βοήθεια πρέπει να δοθεί γρήγορα και αποτελεσματικά δεύτερον για την προστασία των επενδύσεων και τις ξένες άμεσες επενδύσεις πρέπει να υπάρξει σαφέστερος ορισμός των δικαιοδοσιών για να γίνει μια αποσαφήνιση του ποιες είναι οι αποκλειστικές δικαιοδοσίες της Ένωσης και ποιες υπόκεινται στην αναλογικότητα και επικουρικότητα. Είναι πολύ σημαντικό στον τομέα των εμπορικών συμφωνιών και εταιρικών σχέσεων, ιδιαίτερα με τρίτες χώρες, να υπάρξει ένας πραγματικός ορισμός των ιδιωτικών αυτών όταν μιλάμε για εμπορικές συμφωνίες μεικτού χαρακτήρα. Γι' αυτό ο κ. Φερνάντο Ρούες προσβλέπει στη συζήτηση αυτών των θεμάτων σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πρόεδρε, λυπάμαι, αλλά δεν προτιμά σαν λόγο, πρέπει να αυτοσχεδιάσω τώρα. Ήθελα όμως να σας πω ότι είναι ουσιώδες νομίζω αυτό που είπε ο εισηγητής, δηλαδή να δείξουμε πώς, όπως είπε και ο κύριος Βαλέντσα, η επικουρικότητα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, πώς η επικουρικότητα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και πώς είναι απαραίτητη. Βλέπουμε πώς δουλεύει η εξωτερική πολιτική, δεν δουλεύει. Γιατί εκεί υπάρχει πάρα πολλή επικουρικότητα και τα κράτη-μέλη προτιμούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει η εξισορρόπηση. Πολύ δύσκολο. Μεταξύ συγκεντρωτισμού και επικουρικότητας, ιδιαίτερα στη θέματα εμπορικών συμφωνιών. Δεύτερον, για το ISDS, η προστασία των επενδύσεων κλπ. Πρέπει να είναι σαφές ότι ποιες είναι οι δικαιοδοσίες. Αν συζητήσουμε το TTIP και το ISDS στα πλαίσια του TTIP, αυτό πρέπει να το αποσαφηνίσουμε, διότι στα κράτη-μέλη γίνεται συζήτηση, οι εθνικές βουλές πρέπει να επικυρώσουν ή όχι τελικά. Και για μένα δεν είναι σαφές το θέμα. ίσως η έκθεση αυτή να είναι μια ευκαιρία να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα τέλος γιατί δεν σκεφτόμαστε και κάποιο ειδικό είδος επικουρικότητας ειδικό είπε και ο εισηγητής ότι πρέπει οι εκλογές μας να ενδιαφερθούν περισσότερο για την εμπορική πολιτική γιατί δεν κάνουμε πανενοσιακά δημοψηφίσματα για ορισμένους τομείς που ενδιαφέρουν πολύ τους πολίτες. Είναι και αυτό μια δυνατότητα οι εκλογείς να μας πλησιάσουν. Δεν προβλέπεται βέβαια νομικά, αλλά γιατί δεν συζητάμε την πιθανότητα, την ιδέα τουλάχιστον. Και τέλος προσβλέπω στην έκθεση του συγκητή και η σοσιαλιστική ομάδα είναι πρόθυμη να υποστηρίξει ό,τι είναι λογικότερο. Κύριε Σκάρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα των δημοψηφισμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει, θεωρώ, καλύτερος τρόπος να προκληθεί παράλυση στην, ε, στις εργασίες μας. Ίσως όμως έχει κάποιο όφελος. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω. Συνάδελφοι. Το θέμα αυτό το εξετάζω από την πλευρά της Επιτροπής της Νομικών Υποθέσεων εδώ και κάποια χρόνια και φυσικά η επικουρικότητα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το εμπόριο όσο έχει να κάνει με κάποιου άλλου τομεί που δεν είναι στην αποκλειστική ρεμοδιότητα της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνει σεβαστή η επικουρικότητα και η αλλαγικότητα και να γίνει αυτό κατανοητό σε όλα τα θεσμικά όργανα, προκειμένου όλες μας οι δράσεις ε, να έχουν ε, ως σκοπό τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην άσκηση των ε, εξουσιών. Η εμπορική πολιτική των τελευταίων ετών μπορεί να μην έχει τόσο επιρροή στην διαδικασία νομοθεσίας, αλλά είναι σαφές ότι αλλάζει το τοπίο και το μεταβαλλόμενο αυτό το τοπίο θα προαπαιτεί μεγαλύτερη εξέταση των αρχών αυτών. Οι πρωτοβουλίες που συνδέονται με την εμπορική πολιτική και άλλους ε, τομείς, όπως για παράδειγμα η αναφορά των ε, οι εκθέσεις αποκλήφωσης των επιχειρήσεων, δείχνουν με σαφή τρόπο την επικουρικότητα και η επικουρικότητα και η αναλογικότητα θα πρέπει να θεωρούνται εκ των στοιχεία για τη διαμόρφωση της πολιτικής, γιατί ο στόχος της πολιτικών, η στόχη των πολιτικών μπορεί να είναι κοινή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει για τον λόγο αυτό ένα κοινό σκεπτικό και μια κοινή κατανόηση για το πώς επιτυγχάνονται οι σκοποί αυτοί. Γιατί η ευρωπαϊκή δράση δεν είναι πάντα καλύτερη από ότι οι εθνικές δράσεις. Εξετάζοντας λοιπόν το έργο του συναδέλφου μας, του κυρίου Μπορέλη, πρέπει να πω ότι κάποια στοιχεία λαμβάνονται υπόψη. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη δουλειά που έχει κάνει. Ωστόσο, στην παράγραφο 3 πρέπει να επισημάνω ότι πιστεύω ότι κινδυνεύουμε να βγούμε εκτός τροχιάς με το θέμα του ISDS και της προστασίας των επενδυτών. Ίσως δεν είναι εδώ το σημείο να το συζητήσουμε αυτό. Δεν είναι τόσο σχετικό το ζήτημα της έκθεσης. Ένα παράδειγμα να σας δώσω, το οποίο το έχω ελέγξει σε διάφορα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, στο Ενωμένο Βασίλειο υπάρχουν πάνω από 90 ρήτρε ISDS και συμφωνίες από τη δεκαετία του 70 και μετά. Και το Ηνωμένο Βασίλειο ποτέ δεν έχει χάσει κάποια τέτοια υπόθεση σε ό,τι αφορά τον περιορισμό του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου σε ό,τι αφορά την νομοθεσία σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους. Εκεί που υποστηρίζω τον εισηγητή είναι εκεί που αναφέρει την ανάγκη να λαμβάνονται οι αποφάσεις όσο πιο κοντά γίνονται στο πολίτη. Θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή δράση μόνο εφόσον ε, ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει αυτό να γίνεται με, ε, με πλήρη διαβούλευση της κοινωνίας των πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και κλείνοντας να πω, να υπογραμμίσω ένα θέμα ως ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε να ακούσουμε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επικουρικότητα και την αναλογικότητα όχι μόνο στην ε, εμπορική νομοθεσία αλλά και σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες που συνήθισαν προσφάτως, συμφωνίες αλευθέρου εμπορίου. Πρόεδρε, συγγνώμη που ξεπέρασα τα δύο λεπτά. Ναι, όντω λέει ο Πρόεδρος, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα του πόσο γρήγορα μπορεί να εισαχθεί το στοιχείο της επικουρικότητας στην εμπορική πολιτική μία βρετανική μελέτη για θέματα επικουρικότητας. Συμπεράνε ότι όλοι οι τομείς θα πρέπει να επανέλθουν στην εθνική αρμοδιότητα, με μοναδική εξαίρεση το εμπόριο. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν το στοιχείο αυτό, το πώς μπορούμε να εισαγάγουμε την επικουρικότητα στην εμπορική πολιτική. Ίσως να έχει μία απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι από την υπηρεσία για τις διαθεσμικές σχέσεις. Σημειώσαμε πολύ καλά τα σχόλια που έγιναν και όπως είπατε και εσείς ε, ο ίδιος η εμπορική πολιτική είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τομέας σε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι το εκτελεστικό σκέλος η Επιτροπή ε, δεν ε, ακολουθεί στο σύνολο των άλλων πολιτικών την εμπορική πολιτική. Συνεργαζόμαστε με εκπροσώπους των κρατών μελών ε, στενά, αλλά και με εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, τα ερετά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει με το δημοκρατικό έλεγχο. Σημειώσαμε, όπως σας είπα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις και προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία με την Επιτροπή προκειμένου να καταρτήσετε και την έκθεση που προετοιμάζετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπορέλη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συζήτηση. Με ξέπληξε θετικά με ξέπληξαν θετικά οι αξιολογήσεις ε, και κυρίως η αναφορά στο ευρωπαϊκό δημοψήφισμα. Είναι μια πρόκληση και πραγματικά βλέπουμε ότι με τα νέα μέσα, ακόμη και είναι νέα, μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Έτσι λοιπόν, σημειώνω όσα ακούσαμε σήμερα και θα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί του θέματος. Μάλιστα, θα έχουμε λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα την έκθεση στην επόμενη συνεδρία και θα τα συμφωνήσουμε. Και έτσι ολοκληρώνω το σημείο αυτό και περνάμε στο 19 τη ημερήσια διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων για ενδεχόμενη επενδυτική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μιανμάρ. Θα θυμάστε ότι το συζητήσαμε τον Νοέμβριο σε μία ακρόαση. Είδαμε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει. Έως σήμερα δεν υπάρχει συμφωνία από τα κρατημέλη, συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια ορμή στις διαπραγματεύσεις, γι' αυτό και προσβλέπω στις ε, συζητήσεις αυτές. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει πώς έχουν τα πράγματα. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση για το που βρισκόμαστε. Θα έχουμε μια συνέχιση κατόπιν και τις ε, οικρόσεις που ήταν νομίζω πολύ σημαντική. Ο πρώτος γύρος έλαβε χώρα το Φεβρουάριο και όπως είπατε υπήρχε κάποια ορμή. Έχουμε την εντύπωση ότι οι αρχές ε, της ε, Μιανμάρ γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ε, δημιουργηθούν κάποιες ε, ευνοϊκές απαιτήσει επενδύσεων και ε, πραγματικά ήθελα να το καταστήσουν αυτό πραγματικό και για τους Ευρωπαίους επενδυτές. Θέλουν να διαφοροποιήσουν και να μην εξαρτώνται μόνο από συγκεκριμένου επενδυτές. Παρόμοιες συμφωνίες με την Κίνα, την Ινδία, τόσο την Κορέα, την Ιαπωνία... Συνεχίζεται, και καθώς ε, δεν έχουμε διμερή συμφωνία με τα κράτη-μέλη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σημασούμε πρόοδο για πραγματεύσεις αυτές. Συνολικά μπορέσαμε να εξετάσουμε όλο το κείμενο στον πρώτο γύρο. Τώρα θα ήθελα απλώ να σας επισημάνω τα θέματα που νομίζω ότι θα επικεντρωθεί η περισσότερη δουλειά στον επόμενο γύρο το Μάιο. Το ένα είναι οι απαιτήσει επιδόσεων. Αυτή είναι τεχνική γλώσσα για τις απαιτήσει. Ε, να έχουμε περίπτωση χάρη ε, τοπικές ε, συμβάσεις ή απλές απαιτήσει για τους επενδυτές. Επίσης έχουμε απαιτήσει για τη διαφάνεια. Φυσικά υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και είναι δύσκολο να δοθούν έγκαιρες πληροφορίες Μπορεί και αυτό να είναι ένα ζήτημα. Σχόλιο εκτό μικροφώνου, Πρόεδρο. Έχουμε επίση το θέμα τη επίλυση διαφορών, όπου κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για να δούμε πού βρισκόμαστε. Και φυσικά αυτό συμπεριλαμβάνει και το θέμα τη επίλυση διαφορών κράτους επενδυτής, ε, επενδυτή. Άλλος ένας τομέας που μόλις συζητήθηκε σε αυτό τον οίκο. Εμείς ε, επιδιώκουμε πολλές ε, προτάσεις μεταρρυθμίσεων να υλοποιηθούν που έχουμε εφαρμόσει και αλλού, έτσι ώστε να έχουμε έναν ισορροπημένο μηχανισμό επίλυσης διαφορών κράτους επενδυτή. Ε, η πλευρά της BMR γνωρίζει την έννοια αυτή, αλλά ίσως δεν ξέρει το σύγχρονο τρόπο ρύθμισης. Επίσης υπάρχει το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι πολύ θετική η Μιανμάρ σε αυτό το θέμα, σε ό,τι αφορά και τις πτυχές του εργασιακού περιβάλλοντος. Εδώ έχουμε ένα ουσιαστικό κεφάλαιο που δεν ε, είναι οι κανόνες ε, ε, που αφορούν αλλά αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί από την πλευρά της Μιανμάρ για να της Μιανμάρ για να αναλάβουν κάποιες από τις απαιτήσει που τους θέσαμε. Όμως ε, φυσικά δεν λένε ότι δεν θέλουν ε, να υπάρχουν καθόλου κανόνες για την εφόρο ανάπτυξη συμφωνία. Επόμενος γύρος θα είναι στις αρχές Μαΐου. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την επικοδομητική μας συνεργασία για να καταλάβουμε που βρίσκεται η άλλη πλευρά και να κινηθούμε προς ε, μια επιτυχία έκβαση. Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι παράλληλα θα κάνουμε και μία μελέτη αντικτύπου αηφορίας, που νομίζω ότι καλύπτει θέματα σημαντικά και για σας αλλά και για την Κομισιόν σε σχέση με τις ε, πιθανές ε, επιπτώσεις της συμφωνίας ε, στον κοινωνικό τομέα, στον τομέα του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μόνιμος συζητητής, ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν αναφέρθηκε σε κάποια θέματα που ήθελα να τονίσω και εγώ, αλλά θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία, όπως είπε και η Κομισιόν, η Μενμάρη έχει συνάψει κάποιες συμφωνίες μέχρι τώρα. Όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι διαφορετικό το μοντέλο από αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς, το template. Αναφερθήκε το θέμα της ικανότητας Δηλαδή έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν αυτά που ζητάμε εμείς. Έχουν τις δυνατότητες αυτές. Και πώς θα ξέρουμε ε, ποιες είναι οι διαφορετικές από τις εφιστάμενες συμφωνίες με τη Μερμάρ. Τώρα για το κεφάλαιο της αηφόρου ανάπτυξης, ε, το έφερε αυτό η Κομισιόν. Αλλά θέλω να τονίσω κάπως περισσότερο το εξής για το αν απλώς ανησυχούμε για την ικανότητά της να φέρει αποτελέσματα ή αν υπάρχουν κάποιες ε, αντιρρήσεις γιατί ξέρουμε ότι μέχρι τώρα δεν ήταν έτοιμη να σεβαστεί τη σύμβαση του ILO, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Και ξέρετε ότι φυσικά κάποιες ε, πρακτικές ε, στον τομέα της εργασίας ε, συνδέονται. Ίσως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη Μιανμάρ να οδεύσει προς σωστή κατεύθυνση για να έχουμε επιτυχές κεφάλαιο για, το, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, Ακόμη περιμένουμε την Επίτροπο Μάλτρομ να έρθει σε εμά με τη νέα προσέγγιση της Κομισιόν για τις επενδύσεις. Ε, αυτό ποιο αντίκτυπο έχει στη, σας στη δική σας δυνατότητα να διαπραγματευτείτε ε, με την άλλη πλευρά σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο περί επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Στις 7 Μαΐου, νομίζω, θα έχουμε τα νέα στοιχεία που θα μπουν ε, στο κουτί της Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μισό λεπτό να ανοίξει και ο υπολογιστή μου. Στα Ολλανδικά, λοιπόν. Πρόεδρε, θα περιοριστώ στα στοιχεία τα οποία είναι ήδη δημοσιοποιημένα. Καταρχάς, ε, θα ήθελα το ECS να μείνει εκτός της συμφωνίας με τη Μιανμάρ. Η Μιανμάρ προτιμάζει μια ρήτρα ISDS με, με την Παγκοσμία Τράπεζα. και νομίζω ότι αυτό αποτελεί εγγύηση. Αλλά νομίζω ότι και η Μιανμάρ έχει άποψη και θα πρέπει να έχει άποψη για το ISDS. Ξέρετε πόσο δύσκολο και αμφιλεγόμενο το ζήτημα της, ε, του ISDS, της επίλυσης διαφορών κράτους επενδυτού. Ας τους αποφασίσουμε λοιπόν την Μιανμάρ να αποφασίσει η ίδια για την νομοθεσία της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο Μιανμάρ γιατί ουσιαστικά είναι η μη δικτατορία η Μιανμάρ. Το ίμιση των εδρών του Κοινοβουλίου το κατέχουν στρατιωτικοί. Και είναι ξεκάθαρη η πίεση που δέχονται τα μέλη του Κοινοβουλίου να ψηφίσουν προ τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Τον Νοέμβριο έχουν εκλογές στη Μιανμάρα, ελπίζουμε να κάνει ένα βήμα προ μια ολοκληρωμένη δημοκρατία. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο σημείο. Ας μην ε, παραβιαστούμε, γιατί οι συνθήκε είναι πολύ αμφιλεγόμενες και ύποπτες. Γιατί να μην ε, διακόψουμε τις διαπραγματεύσεις ε, τις οποίες να τι διαπραγματεύσει και να τι ξαναξεκινήσουμε μετά τι εκλογέ. Δεν είναι ρητορικό το ερώτημα αυτό. Θέλω απάντηση. Τέλο. Ε, από ό,τι καταλάβα, ο Επίτροπο μίλησε με εκπροσώπου 23 ε, κοινωνικών οργανώσεων που ήταν κατά τη εμπορική συμφωνία. Ε, ποια ήταν τα αποτελέσματα των συζητήσεων και αυτό τροποποίησε καθόλου την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Σύντομη. Για τις διαπραγματεύσεις τον Μάιο, τι προβλέπετε, τι ακριβώς θα συζητηθεί. Δεύτερον, αναφέρατε ήδη τις απαιτήσει αποδοτικότητας, αλλά τι ισχύει και γι' αυτό, αφού είναι θέμα προστασίας επενδύσεων και όχι πρόσβαση στις αγορές. Επομένως νομίζω ότι η Κομισιόν δεν πρέπει να συζητήσει τις χαρακτηριστικές αποδοτικότητες γιατί η Μιανμάρ είναι φτωχή χώρα. και πρέπει ορισμένη ενωτμήμα της έρευνας να γίνει επιτόπου και να μην απαγορεύονται οι μεταφορές τεχνολογίας. Πρέπει να κάνει ακόμα πολύ δρόμο η χώρα για να αναπτυχθεί. Επίσης γνωρίζουμε ότι στη Μιανμάρ υπάρχει μεγάλη αντίθεση σε αυτά τα κριτήρια αποδοτικότητας. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί πρέπει να συμπεριληφθούν και θα μπορεί η Μιανμάρ να επιχορηγεί εγχώριους επενδυτάς. Επίσης μιλήσατε λίγο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εμείς δεν νομίζουμε ότι είναι σωστό να συμπεριληφθεί το ISDS στη συμφωνία με τη Μιανμάρ. Γιατί πρέπει ακόμη να διορθωθούν και να διευθετηθούν πολλά στη Μιανμάρ. Ενώ η ISDS περιορίζει τέτοιες δυνατότητες όπως ξέρουμε και από τις συζητήσεις μας επ' αυτού. Όσο για τις αξιολογήσεις αντικτύπου, και ο αρμόδιος επίτροπος για το εμπόριο είπε ότι ο ειδικό συζητητής του ΟΗΕ δέχεται ορισμένες εξαιρέσεις. Θα δεχτείτε λοιπόν αυτά που είπε και ο ειδικό εκπρόσωπος του ΟΗΕ. για μια αναπτυσσόμενη χώρα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω αρχίζοντας με το ερώτημα δυνατοτήτων και βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα από τα κύρια θέματα είναι βέβαια η σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που δεν έχει επικυρωθεί από όλους και με επιχείρημα ότι προσπαθούν να τα εφαρμόσουν αυτά μέσω τοπικής νομοθεσίας αλλά όχι ως πλήρη εφαρμογή της σύμβασης. Κανείς δεν ξέρει πόση αντίσταση υπάρχει από το σύστημα. Εμείς βλέπουμε την πρόσωψη μόνο. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους που θέλουν να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα και δεν θέλουν να υπογράψουν κάτι που δεν θα μπορούν να το εφαρμόσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, πολύ σκληρά όμως, πάρα πολύ σκληρά. Γιατί θέλουμε να δοθεί αξιόπιστη απάντηση σε αυτό το πρόβλημα στη Μιανμάρ. Όσο για τη σύμβαση του αγελό δεν συνδέεται απαραίτητα θα μπορούσαμε και με τον τρίτο πυλώνα να κάνουμε ορισμένες δαπάνες για την εφαρμογή των εργατικών νόμων, εργασιακών νόμων. Για μας η ύπαρξη ενός αναπτυξιακού προτύπου στην ή για την Μιανμάρ είναι ουσιώδης. για το νέο ISDS νομίζουμε ότι γνωστοποιούμε σε όλους μας τους εταίρους περί τίνος πρόκειται. Τους λέμε ότι αν καταλήξουμε σε μία λογική μεταρρύθμιση τότε μπορεί να επιτραπεί κάποια αλλαγούλα. Μετά υπάρχει το θέμα που έθεσαν η κυρία Βίμερ και η κυρία Κέλλερ να μην συμπεριληφθεί καθόλου το ISDS. Εδώ το μόνο που θέλω να πω είναι το εξή. Πρώτον, η Μιανμάρα επιτρέπει σε πολλούς τοπικούς παράγοντες προστασία και είναι δύσκολο να εξηγήσουμε γιατί εμείς δεν το θέλουμε αλλά επειδή πρόκειται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, επακρόθεσμες, πρέπει να δούμε και τι μπορεί να γίνει μετά από καινούργιες εκλογές ας πούμε. Αν θέλουμε να εφαρμοστούν τα κριτήρια αποδοτικότητας, αυτό είναι συζητήσιμο για τις αναπτυσσόμενες χώρες μερικές φορές είναι καλά αυτά τα θέματα θετικά αλλά θα δούμε τι έχουν να πούν και οι άλλοι διαπραγματευτές οι εταίροι μας οτιδήποτε, οποιοδήποτε εθνικό μέτρο μπορεί να είναι αποδοτικό, το συζητάμε αλλά επίσης μπορούμε να είμαστε και ελαστικοί ώστε να μην ακυρώσουμε αυτά που έχουν ήδη συμφωνήσει με τους Ιάπωνες και ό,τι άλλο έχει ήδη αναλάβει ως δέσμευση η Μιανμάρ. για να μην είναι λιγότερη προστασία των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις δεν είναι θέμα. Δεν θα δεχτούμε καμία επιχορήγηση που θα ζητήσει η κυβέρνηση της Μιανμάρ. Όσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το SIA, θα ήθελα να επαναλάβω ότι οι αξιολογήσεις αντικτύπου στοχεύουν, ε, δίνονται από κάποιον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που κοιτάζει όλα τα θέματα. Θα δούμε τι έχουν να πούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλοι οργανισμοί όπως πρακτορία του ΟΗΕ. Μια ερώτηση διευκρινιστική. Είπατε ότι η Μιανμάρα έχει συνάψει τρεις ε, ε, συμφωνίες, ε, έχει υπογράψει τρεις συμβάσεις της ΔΟΕ επί των οκτώ. Μετά από πόσε ε, τέτοιες πιστεύετε ότι, ε, πόσες τέτοιες πιστεύετε ότι πρέπει να υπογραφούν για να πούμε ότι γίνεται σεβαστό το εργατικό δίκαιο. Κομισιόν, κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλούς ε, που έχουν προσυπογράψει τις συμβάσεις ε, της ΔΟΕ. Αλλά ποια είναι η διαφορά επιτόπου, αυτό πρέπει να δούμε. Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να υπογράψει η χώρα την εφαρμογή επί της ουσίας. Δηλαδή να δούμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτό, πώς το κάνετε και εδώ επισέρχεται και εθνική νομοθεσία. Αλλά στις διεθνείς σχέσεις δεν, δεν βασιζόμαστε στη ΔΟΕ. Έχουμε μία πρόβλεψη στη συμφωνία ότι εμείς θα παρακολουθούμε με τα δικά μας μέσα την εφαρμογή της αηφόρου ανάπτυξης. Ε, γιατί το να υπογράφονται πολλά χαρτιά τελικά δεν μας οδηγεί στο να έχουμε ένα μέσο για να ελέγχουμε τι συμβαίνει. Γι' αυτό δίνεται και πολύ μεγάλη προσοχή στην παρακολούθηση. Δεν λέμε ότι αρκούν οι τρεις. Κάποιες χώρες έχουν περισσότερες ή λιγότερες. Οι ΗΠΑ αναφέρθηκαν πολλάκις. Ακριβώς ε, κατάλαβα τι ακριβώ προσπαθείτε να πείτε. Το ξέρω, η απάντηση είναι η ίδια. Προσπαθούμε να υπογράψουν ε, οι χώρες επί της ουσίας ε, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το λαό επιτόπου, πέρα από το θέμα της κύρωσης Φυσικά μια σύμβαση διεθνούς δικαίου είναι πολύ καλύτερη από μια διμερή συμφωνία. Πρόεδρος, νομίζω ότι σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε πολλές ε, συζητήσεις την επόμενη φορά. Θέλω ο να πει κάτι, όχι. Ωραία, ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε το σημείο 19 και θα περάσουμε στο σημείο 20. Αυτό θα γίνει και κλεισμένον το θυρών, όπως και το επόμενο σημείο η συνεδρίαση των συντονιστών. Επομένως, μόνο τα μέλη της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, οι βοηθοί, οι πολιτικές ομάδες, η νομική υπηρεσία, το πολιτικό τμήμα και η γραμματεία της ΣΥΝΤΑ επιτρέπεται να μείνουν στην αίθουσα. Οι άλλοι παρακαλούν να αποχωρήσουν.